I think we can start. Please sit down. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer letzten TRAN-Ausschusssitzung. Σας ε, καλωσορίζω στην τελευταία μας ε, συνεδρίαση για φέτος της Επιτροπής ε, ΤΡΑΝ, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, και ε, περνάω στο πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης, ε, ε, έγκριση λοιπόν του σχεδίου ημερήσιας διάταξης, αλλά όπως ε, γνωρίζετε έχει αναβληθεί ψηφοφορία σε ό,τι αφορά το συνδρομικό πακέτο, αλλά κατά λοιπά νομίζω πως μπορεί να εγκριθεί μέσα σε διάταξη. Ε, και θα, σας, θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην Αλποφιλίψα για, για την αεροπορία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, να δώσω κάποιες διευκρινήσεις ε, γιατί αποστάλησαν κάποια email κατά τις τελευταίες τρεις ημέρες, οπότε θα ήθελα λίγο να σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως γνωρίζετε, η δική μου πρόθεση με τη σύμφωνη γνώμη των ε, σχεδόν εισηγητών ήταν να εκπονήσουμε μία σύντομη και περιεκτική έκθεση ως προς το τι θεωρούμε πως ε, πρέπει να αποτελέσει ζήτημα προτεραιότητας αλλά και τι, ε, ποια είναι τα κενά του σχετικού πακέτου. Και χαίρομαι και να το πω αυτό ευθύ εξ αρχή ότι καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία με του σκιώδει συζητητέ. Γιατί καταφέραμε πραγματικά να εργαστούμε με ταχύτητα και καταλήξαμε σε ένα κείμενο το οποίο καλύπτει όλα τα ε, ζητήματα που θέλαμε με έτοιμον παραγραφό το κάθε ένα από αυτά Οπότε δεν έχουν προκύψει ζητήματα ως προς τις επιμέρους προτάσεις που έγιναν από τους διάφορους συναδέλφους. Το επιτύχαμε λοιπόν αυτό και κάτι ακόμα που έκανα και το οποίο πραγματικά συμμορφώνεται με το καταστατικό μας ε, εδώ, το τονίζω δηλαδή, και δεν βασίστηκα εδώ στα όσα μου είπε η γραμματεία, αλλά διάβασα εγώ ο ίδιος τους κανόνε του καταστατικού, είναι λοιπόν να καταρτήσουμε μία ε, γνωμοδότηση ε, που αποτελείται από 35 ε, διαφορετικές παραγράφους, δηλαδή τον ίδιο ακριβώ αριθμό παραγράφων με αυτέ που συμπεριλαμβάνονταν στην έκθεση. Δεν ξέρω ε, κατά πόσο όλοι σας συμφωνείτε με το να έχουμε μια σύντομη έκθεση από ε, κοινό με τους εστιώδεις, αλλά ε, ουσιαστικά μια χνομοδότηση η οποία είναι τόσο σύντομη δεν ανταποκρίνεται στον ίδιο βαθμό στο περιεχόμενο της έκθεσης παρόλα αυτά και τα δύο αυτά ε, έγγραφα καλύπτουν τα ζητήματα ε, των ε, αρμοδιοτήτων, κοινών αρμοδιοτήτων και αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της δικής μας Επιτροπής Τραν. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με το νέο έγγραφο είναι να εκπονήσουμε ένα σύντομο κείμενο το οποίο εξακολουθεί να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είχαν συζητηθεί ε, στο επίπεδο των εισηγητών προκειμένου να αντιμετωπιστεί στην Επιτροπή. Και νομίζω πως σωματικά θα συγκεντρώσει με ισχυρή πλειοψηφία αυτό το κείμενο. Τώρα, στην ιδανική περίπτωση, Κάποιοι συνάδελφοι εδώ ουσιαστικά δεν θα υπέβαλαν τροπολογίε οι οποίε δεν αποτελούν τόσο άλλο δική μα αρμοδιότητα, αλλά αρμοδιότητα τη Επιτροπή για την Απασχόληση. Και βέβαια ε, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Τώρα, ε, χρειαστεί να ψηφίσουμε από αυτού του εγγράφου, ναι θα χρειαστεί, γιατί νομίζω πω αναφέρεται αυτό με σαφήνα και στο καταστατικό μα ότι δηλαδή πρόκειται καταρχήν για αρμοδιότητα του ΕΣΥΤΗ και από εκεί και μετά γίνεται ψηφοφορία. Άρα δηλαδή η Επιτροπή Απασχόλησης μπορεί να πάρει την γνωμοδότησή της και να την επανυποβάλει στην Ολομέλεια. Αν εμείς δεν επιθυμούμε να την εξετάσουμε εδώ οπότε. Χωρί να θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γραμματεία για τη συνεργασία που είχαμε ε, και να πω: Έχουμε τηρήσει όλους τους σχετικού ε, κανόνε του καταστατικού. Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε μια πολύ καλή ποιότητα στη δική μας έκθεση, ούτως ώστε να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα και προκειμένου να βρίσκεται στα χέρια της Επιτροπής έγκαιρος, ούτως ώστε να, ε, δηλαδή προτού υποβάλει σχετικές προτάσεις της για μια σειρά αποζητήματα η Επιτροπή στις αρχές του επόμενου χρόνου. Ε, αν δεν ακολουθήσουμε ε, τα όσα προτείνω εγώ θα καθυστερήσουμε ακόμα περισσότερο σχέση δηλαδή με την πληροφορία στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Οπότε αυτό που λέω εγώ είναι να ακολουθήσουμε τους κανόνες του, ε, του καταστατικού, ώστε τα ζητήματα που είναι μεικτής αρμοδιότητας και αποκλειστικής αρμοδιότητας της δικής μας Επιτροπής ΕΤΡΑΝ να ψηφιστούν εδώ στο δικό μας επίπεδο της Επιτροπής. Ασχέτως δηλαδή θα γίνει με τα υπόλοιπα ζητήματα της Επιτροπής Απασχόλησης. Οπότε, ε, αν θα ήταν δυνατό και σας παρακαλώ να το κάνουμε αυτό, ε, Πρόεδρε, να υπάρξει μια πολύ σύντομη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ε, εδώ, επιτροπή Επιτροπής δηλαδή Τραν, προτού ε, περάσει το σχετικό ζήτημα για ψηφοφορία στην Ολομέλεια, αν αυτό είναι δυνατόν. Θα πρέπει να αναργονίσουμε τα όσα έχουμε καταφέρει εδώ και να πούμε ότι υπήρξε ούτω ή άλλω σε σχέση με αυτέ τι απόψει έχουμε στο έγγραφό μας ισχυρή υποστήριξη από όλε τις πολιτικές ομάδες. Και ταυτόχρονα σεβαστήκαμε πλήρως τους κανόνες του καταστατικού. Θα ήθελα στο μέλλον να αποφύγουμε τέτοιου είδου καταστάσεις. Και να ζητούμε δηλαδή ότι όταν υπάρχει μία έκθεση την οποία εμείς ε, προτείνουμε και περιλαμβάνει 35 σημεία, 35 παραγράφους, να μην λαμβάνουμε μια γνωμοδότηση από μια άλλη επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει τον ίδιο αριθμό παραγράφων ή σημείων. Γιατί κάτι τέτοιο μόνο δυσκολεύει τις ε, ε, εργασίες μας. Πρόεδρος. Πράγματι, αναφέρθηκε αυτό, ε, ότι δηλαδή είχαν ε, η γνωμοδότηση και η έκθεση το ίδιο μέγεθο, ένα το ίδιο μακροσκελή, αλλά από εκεί και μετά τίθεται και το ερώτημα του τι συμβαίνει σε περίπτωση αποκλειστική αμοδιότητα μια συγκεκριμένη επιτροπή. Σε πάση περιπτώσει, ε, θα συζητήσουμε τώρα στην συνάντηση των συντονιστών που θα ακολουθήσει το αν θα γίνει μια ξεχωριστή ψηφοφορία την ερχόμενη εβδομάδα τη Επιτροπή μα. Δεν θα ανοίξω το λόγο. Ε, δεν θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου για συζήτηση. Δεν θα κάνουμε συζήτηση τώρα. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στι ψηφοφορίε. Και περνάω λοιπόν στο σημείο για την εφοδιαστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πολυτραπικέ μεταφορές στου νέου διαδρόμου διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Ινέσα Σαγέλα Σάντερ είναι η συγγήτριά μα. Οπότε, ας ελέγξουμε καταρχήν. Ας ελέγξουμε λοιπόν, να ψηφίσουμε όλοι δοκιμαστικά. Δεν έχετε κάρτα σαν Το σημειώνουμε. Οπότε θα μου κάνετε ένα νόημα και θα σας κοιτάω πάντα για τις ψηφοφορίες. Ναι. Ωραία. Όλα καλά λοιπόν, τουλάχιστον προς το παρόν. Παραγράφος 1, λοιπόν, τοπολογία 25. Αναφερόμαστε στο σχέδιο έκθεση για την εφοδιαστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μεταφορέ, έτσι. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία για την τροπολογία 25. Πέραση της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 22 κατά. Άρα απορρίπτεται. 22 γιατί η Τζάκη Φώστερ ψήφισε κατά και η Τζάκη Φώστερ δεν έχει κάρτα τη σήμερα εδώ. Καλώς, το διευκρινίσαμε. 26 τώρα τροπολογία ψήφι περ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε λοιπόν τη 49 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας 30 Σε 5, 13 κατά εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2α υπέρ κατά αποχές εκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 58 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. 22 ψήφοι υπέρ. 21 ψήφοι κατά. Εκρίνεται λοιπόν. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται. 60. Με την προφορική τροπολογία. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική, οπότε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά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 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 22 υπέρ 23 κατά καμία αποχή οπότε απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 140 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 150 ηλεκτρονικά Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 21, 21 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά, 3 αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. ...145 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. NV21 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε την NB21, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 23 ψήφοι υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται λοιπόν. NB22 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV9 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την NBNA ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία, 22 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, 5 αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές 155 να ελέγξουμε. τη ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 25 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, 3 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. NV3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. NV7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. NV13 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NB17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NB19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 202 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε την 202. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας, 22 ψήφοι υπέρ, 23 ψήφοι κατά απορρίπτεται. 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική, α όχι, να ελέγξουμε την τροπολογία 203 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας, 32 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται λοιπόν. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 12 λοιπόν ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέραση ψηφοφορίας 20 ψήφοι υπέρ, 25 ψήφοι κατά, 0 αποχές απορρίπτεται, 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβη 18 υπέρ τμήματική ψηφοφορία τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τοπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τροπολογία 2 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας 21 ψήφι υπέρ, 21 ψήφι κατά, 3 αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε και την τροπολογία 3 λοιπόν, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21 ψήφι υπέρ, 21 ψήφι κατά, 3 αγωχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την 8 δεν ψηφίζουμε οπότε περνάμε στο κόλπο τελική ψηφοφορία λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το σύνολο πέραση της ψηφοφορίας 40 ψήφοι υπέρ 4 ψήφοι κατά καμία αποχή τα συγχαρητήριά μας στην Σύγκριση. Α, όχι, 41 ψήφοι πέρα, διορθώνει ο πρόεδρος. Herzlichen Glückwunsch. Συγχαρητήρια. Which one? That is... So, wir kommen jetzt zur nächsten Abstimmung. Να περάσουμε στην επόμενη ε, ψηφοφορία για το πακέτο των συνδρομικών μεταφορών. Έκθεση Wim van den Kamp. Σχέδιο συστάσεων σε δεύτερη ανάγνωση σε ό,τι αφορά την ε, του κανονισμού, την έξοδο του κανονισμού για το άνοιγμα της αγοράς ε, για τις μεταφορές αυτές. Για το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών συνδεδρομικών μεταφορών. Μάλιστα. Έτοιμοι. Έκθεση Φαντεντ Κάμπ. Τροπολογία 1 και 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Η τραπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 5. Ένταρξη. Πέρας. 19 υπέρ, 26 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. Η 6 υπέρ. Ή 6 και 7 μάλλον μαζί. Υπέρ. Από κοινό. Από κοινό. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Η 3 και η 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινονται. Τελική ψηφοφορία. Έναρξη παρακαλώ ψηφοφορίας με ονομαστική κλίση. Πέρας. 30 υπέρ, 15 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια προς τον κύριο Βιν Κάμπ. Εγκρίθηκε η έκθεση του. Και τώρα, έκθεση σας όλοι. Για την τροπολογία 1 και 2 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 9. Έλεγχος. Για την 3 έως 8. Όχι, όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Ω, τώρα θα ελέγξουμε. Έναρξη, λέει ο πρόεδρος. Πέρας. 25 υπέρ 20 κατά. Καμία αποχή εγκρίνονται. Η εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Τελική ψηφοφορία για την έκθεση σας όλοι. Έναρξη. Πέρας. 31 ψήφοι υπέρ, 14 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Jetzt der Έκθεση Kielönen. Διευθέτηση λογαριασμών των συνδρομικών επιχειρήσεων. Τελική ψηφοφορία. Μία και μόνη. Με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Πέρασε. 42 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Τεράστια πλειοψηφία. Συντριπτική συγχαρητήρια. Jetzt kommt der Bericht von Karamadeli. Wir kommen jetzt zum Bericht. Να περάσουμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Καριμαντέλη για την αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πρωτού περάσουμε στις ψηφοφορίες, θα ήθελα για τα πρακτικά να αναφέρω το εξή. Οι τελευταίες τροπολογίες ε, κατέφθασαν ε, και συμφωνήθησαν την Παρασκευή το βράδυ και οι πιο πολλές γραμματείες ε, τις ε, έλαβαν ουσιαστικά σήμερα το πρωί. Εμείς ε, λοιπόν ως σοσιαλιστές θα μάθαμε αυτά σήμερα το πρωί και ως εκ τούτου δεν μπορέσαμε να εκτάξουμε σε μεγάλη λεπτομέρεια τις τροπολογίες αυτές και γι' αυτό λοιπόν να συμφωνήσουμε στο μέλλον να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο για τις συμβαστικές τροπολογίες, να έχουμε και εμείς το χρόνο μας να τα κοιτάξουμε. Δεν ε, καταφέραμε λοιπόν να τι κοιτάξουμε όσο θα θέλαμε και αυτό δεν είναι ιδανικό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος και έτσι είναι τα πράγματα. Καλύτερα ποιότητα παρά ταχύτητα. Μπορεί να γίνει και αναβολή. Δύσκολο βέβαια, αλλά παρ' αυτά το αποδεχτήκατε να ψηφίσουμε. Στο μέλλον όμως να φροντίσουμε να λαμβάνουμε τις τροπολογίες, ε, όχι ε, Παρασκευή βράδυ, πιο εγκαίρος και Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου, ως γνωστόν. Έκθεση Καρυμαντέλη τώρα. Τροπολογία 101, υπέρ. Κατά. Μα δεν σηκώσατε τα χέρια σα υπέρ, λέω. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 102 υπέρ. Θέλετε έλεγχος για την 101. Να γίνει. Εντάξει λοιπόν. Έναρξη. Εδώ έλεγξαμε άλλα κι άλλα. Πέρα για την 101. 37 η ψήφη υπέρ, 8 κατά, καμία αποχή. Δεν ήταν ωραία το αποτέλεσμα, εγκρίθηκε. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίθηκε. 103 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 103 παρακαλώ. Πέρας. 26 ψήφοι υπέρ, 18 κατά, μία αποχή εγκρίθηκε. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 106 υπέρ κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε παρακαλώ, ελέγχουμε την 106. Πέρασε. Α, τι θα κάνετε, απέχετε. 22 υπέρ, 23 ε, κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 107. Ας ελέγξουμε. Πέρασε. 22 υπέρ, 23 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. Ευχαριστώ. Αλλά σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. 108 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 108. Πέρας. 22 υπέρ, 22 κατά, μία αποχή απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε πολλές σελίδες. 116 υπέρ. Να περιμένω, να περιμένω λίγο. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 13. Έναρξη. Πέρας. 19 υπέρ, 22 κατά, 3 αποχές απορρίπτεται. 117, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Έλεγχος συζητείται για την 144. Έναρξη. Πέρας. 11 υπέρ, 32 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας αλλάξουμε παρακαλώ τον 21. Έναρξη. Πέρας. 21 ψήφοι υπέρ, 21 κατά, μισοψηφία απορρίπτεται, 176 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ για την 28. Έναρξη. Πέρας. 23 υπέρ, 21 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 182 και 183 μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος παρακαλώ για την 184. Πέρασε. 25 υπέρ, 19 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε. Την 194 υπέρ. Συγγνώμη, έναρξη. Πέρασε. Τζέκι. 27 υπέρ, 17 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 34. Α, όχι, καταπληκτή, 198 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 201 η 198 α, έλεγχος. Έναρξη παρακαλώ. Πέρας. 15 υπέρ 29 κατά καμία αποχή απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 201. Έναρξη. Πέρας. 25 υπέρ 19 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ τι γίνεται με την 219. Έναρξη. Πέρας. κάνει υπέρ, 25 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. 222 και 223 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας αλλάξουμε 225. Έναρξη. Πέρας. 31 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 40 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε. Ελέγχουμε παρακαλώ την 40. Πέρας. 30 υπέρ 14 κατά. Καμία αποχή εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε και την 229 παρακαλώ έναρξη. 20 υπέρ, 22 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 231 και 232 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την 236. Έναρξη. Πέρας. 22, υπέρ, 22 κατά. Μισοψηφία, καμία αποχή, απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 235. Α, όχι καταπίπτει. Η 42 τότε, υπέρ. Κατά. Έλεγχος για τη 42. Έναρξη. Πέρας. 20 είναι υπέρ, 15 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 241 και 41 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 242 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ τη 43. Έναρξη. Πέρας. 21 υπέρ, 23 κατά, καμία απόχη, απορρίπτεται. Η 256 υπέρ. 46, συγγνώμη, υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 247 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 268 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 και 271 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. 44 και 271. Παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Τρίτα μία ψήφι υπέρ, 13 κατά καμία αποχή εγκρίνεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε και τη 272 παρακαλώ. Έναρξη. Πέρας. 26 υπέρ, 18 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 275 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 277 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε τι γίνεται με την 6 παρακαλώ. Έναρξη. Πέρας. 24 υπέρ 19 κατά καμία αποχή εγκρίνεται. Η 297 και 298 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 300 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 303 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 304 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 324. Έναρξη. Πέρας. 28 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. 319 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 320 Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 321 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 322 και 323 υπέρ. Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε. 322 και 323 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρασε. 19 υπέρ, 21 κατά, 2 αποχές απορρίπτεται. 324 παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 325 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 326 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 327 και 328 υπέρ, κατά Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 52 παρακαλώ. Έναρξη. Πέρας. 23 υπέρ, 19 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Η 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 330 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 330 παρακαλώ. Πέρας. 20, 19 μάλλον υπέρ, 21 κατά καμία αποχή. Απορρίπτεται. 335 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 337 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.41 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 3.44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 3.46 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε την 56. Έναρξη. Πέρας. 21 ψήφι, υπέρ 19 κατά καμία απόχη, εγκρίνεται. Ή 57 υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω τίποτα. Για την 57 λέω, υπέρ. Κατά. Εποχές, ας ελέγξουμε την 57 και ηλεκτρονικά. 26 υπέρ, 16 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. 58 και 351 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Η 353 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 357 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 359 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 358 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 360 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 360 έναρξη. Πέρασε. 24 υπέρ 19 κατά καμία αποχή εγκρίνεται. 364 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 367 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 372 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 374 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 376 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 393 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε. Την 34 παρακαλώ. Έναρξη. 26 υπέρ, 17 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 36 παρακαλώ. Έναρξη. Πέρας. 20 υπέρ, 23 κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. Η 60 υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε την 60 παρακαλώ. Έναρξη. Πέρασε. 20 υπέρ, 23 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. Η 399 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 400 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 434. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 435 υπέρ. Έλεγχος για την 64. Εντάξει. Για την 64 λοιπόν ψηφίζουμε. Πέρας. 13 υπέρ, 27 κατά, 2 αποχές και αυτό δεν ήταν οριακό. 435 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 436 υπέρ. Κατά. Αποχές Ας αλλάξουμε την 436 παρακαλώ έναρξη. Πέρασε. 25 υπέρ 18 κατά καμία αποχή εγκρίνεται. 438 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 68 παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Πέρας. 18 υπέρ, 25 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. 441 ε, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 445 υπέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.49 και 4.50. 450 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 455 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 476 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 477 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 479 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 480 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 491 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4.94 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος για την 4.94. Πέρας. 23 υπέρ, 20 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. 4,95 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 495. Πέρας. 35 υπέρ 8 κατά καμία αποχή εγκρίνεται. 502 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 514 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 514. 17 υπέρ, 26 κατά, καμία αποχή, απορρίπτεται. 515 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 516 υπέρ. Κατά. Αποχές, ας ελέγξουμε και την 516. Πέρασε. 28 υπέρ, 15 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. 518 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 520 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 522 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 523 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 527 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 525 υπέρ κατά εγκρίνεται. 533. Α, α, αποσύρθηκε. 534 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 535 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 536 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 537 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 541 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 541. Έναρξη. Και πέρας. 17 υπέρ, 26 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. 542 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε τη 2. 2. Πέρασε. 20 υπέρ, 22 κατά, καμία αποχή απορρίπτεται. Η 3 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 72. 72. Ναι, σας ευχαριστώ. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 73. Έναρξη. Πέρας. 14 υπέρ, 29 κατά καμία αποχή απορρίπτεται. Η 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 83. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Να ελέγξουμε την τροπολογία υπερθμών 9. Ψηφίζουμε. Περάς. 21 υπέρ, 21 κατά, καμία αποχή, απορρίπτεται σε ισοψηφία. 85 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για τη 10. Έναρξη. Πέρας. 19 υπέρ, 22 κατά καμία αποχή. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν φαίνεται. 99 παρακαλώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ένταξη. Και πέρασε. 21 υπέρ, 21 εκατά. Καμία αποχή απορρίπτεται. Με τροπολογία 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μάλιστα. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστικά. Α, όχι κανονικά. Έναρξη. Πέρας. 34 υπέρ, 6 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια στην κυρία Ντελή. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι να προσέλθει η Επίτροπος. Μπορείτε να πιείτε ένα καφέ έτσι. Ναι. I think we can start. Please take a seat. Νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ich komme zu unserem nächsten Tagesordnung. Περνάω στο επόμενο σημείο της μέσης διαταξής μας, ε, δηλαδή τη συζήτηση με την Επίτροπο μεταφορών, Βιολέτα ε, Μπούλτς. Ε, σας ε, καλωσορίζω λοιπόν με μεγάλη μου χαρά για μία ακόμα φορά εδώ στην Επιτροπή μας. Η Επίτροπος Ζαμπούλης θα μας παρουσιάσει καταρχήν το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το έτο 2017 και στη συνέχεια θα προβούμε σε μια γενική συζήτηση σε ό,τι αφορά την κατάσταση τη ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, γιατί βέβαια υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε πιο κοντά στου στόχου μα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνενωθεί ακόμα καλύτερα, θα πρέπει να διατηρηθούν αλλά και να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία και να προστατεύσουμε ε, το περιβάλλον. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που πρέπει να κάνουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να τα κάνουμε πολλά πράγματα τα ίδια έχουμε καταφέρει, δηλαδή μεταρρύθμιση των συνδρομικών μεταφορών, ο κανονισμό ε, για του λιμένου ή και ο κανονισμό σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό Ασφάλεια τη Αεροπορία, την ΕΑΣΑ δηλαδή, και την νομοθεσία σε την ασφάλεια στη θάλασσα. Αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία που λείπουν ακόμα, όπω για παράδειγμα ε, το πακέτο για τι οδικέ μεταφορέ, το οποίο έχει ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό, ο κανονισμό 868 σε ό,τι αφορά την αεροπονιστικότητα τη αεροπορία, αλλά και ο κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών στι αεροδρομικέ ε, μεταφορέ. Και υπάρχει βέβαια και το ζήτημα της εφαρμογής στην πράξη ε, των αποφάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας της ΕΚΑΟ σε ό,τι αφορά ε, την ε, μείωση των εκπομπών. Χαίρομαι λοιπόν που είστε σήμερα μαζί μας εδώ κυρία Μπούλκ και σας δίνω το λόγο για να κάνετε την παρουσίαση σας. Mr. Chair. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι έκτη φορά το τελευταίο χρόνο που έρχομαι εδώ. Σε συνεδρία στη δική σας ή των συντονιστών. Πέρα όλων των διμερών, επαφών, δείπνων και οτιδήποτε άλλο έχουμε κάνει. Οπότε με χαρά λοιπόν είμαι εδώ μαζί σας. Ιδιαίτερα για να σας μιλήσω για σημαντικά θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν θετικά το 2017. Ζητήσατε να σας πω πολλά και στο τέλος συζήτηση σήμερα θα δείτε ότι θα σας πω όντως πολλά. Πριν προχωρήσω όμως να σας πω χρόνια πολλά. Ισμαν Χέρτου, χρόνια πολλά. I must excuse, I didn't do Α, εγώ ζητώ συγγνώμη, δεν το έκανα. Δεν είπα χρόνια πολλά κι εγώ. December gives quite... Ο Δεκέμβρης είναι ευκαιρία απολογισμού του έτους Πολλά λοιπόν έγινε το 16. Λίγα από αυτά. Σημαντικοί φάκελοι ολοκληρώσαμε δύσκολες διαπραγματεύσει για το σιδηρόδρομο και τους λιμένες και συγχαρητήρια για τη σημερινή ψηφορία γιατί πραγματικά με στηρίζει πολύ και μου δίνει εμπιστοσύνη όσον αφορά τη φάση εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός λοιπόν από το τέταρτο πακέτο και τις λιμενικές υπηρεσίες όπως έλεγα Επίσης, βασίζομαι πάνω σας για να υιοθετήσουμε συγκεκριμένα πράγματα στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα, όπως η, η έναξη διαπραγματεύσεων με σημαντικούς εταίρους στον τομέα της αεροπλοείας. Σήμερα πάντως θα εστιάσω στο μέλλον και θα αναφέρω σύντομα το ότι θα βρούμε μπροστά μας το 2017. CITS και στρατηγική. Καταρχάς, η νέα πρωτοβουλία που θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι η στρατηγική που εθετήσαμε σε επίπεδο Κομισιόν την περασμένη Τετάρτη. Δεν είναι μυστικό ότι θα ήθελα τώρα να δω τα πρώτα συνδεδεμένα οχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους μέχρι το 19. Αυτή λοιπόν η στρατηγική θα μας βοηθήσει να τα πετύχουμε αυτά είναι ουσιώδη για να διασφαλίσουμε ότι η υποδομή μεταφορών και τα οχήματα θα αρχίσουν να συνεργάζονται μέχρι το 2019. Αυτό λοιπόν θα κάνει τους δρόμους μας ασφαλέστερους, θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και θα μας βοηθήσει να ενσωματώσουμε στα συστήματα μεταφορών μας τα αυτοματοποιημένα οχήματα κύριοι στόχοι στρατηγική είναι καταρχά να αποφύγουμε ένα, μια κατακαιρματισμένη εσωτερική ενιαία αγορά, να καθορίσουμε προτεραιότητε και στόχου, να χρησιμοποιήσουμε ένα μείγμα τεχνολογιών και επικοινωνιών, να αντιμετωπίσουμε θέματα προστασία δεδομένων και ασφάλεια και να αναπτύξουμε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, όπω βεβαίω και να συνεργαστούμε σε διεθνέ επίπεδο. Αυτή λοιπόν η στρατηγική διασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και για ιδιώτε αλλά και για το δημόσιο ω επενδυτέ. Επίση, ασχολείται με το θέμα τη διαθεσιμότητα κονδυλίων για προγράμματα έρευνα και ανάπτυξη για διεθνούς συνεργασίες, όπως επίπεδο G7 α πούμε. Δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξή. Η στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Τον περασμένο Σεπτέμβρη σα παρουσίασα τη νέα μα στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Κάποιοι με ρωτήσατε πότε θα τα εφαρμόσουμε όμω όλα αυτά. Ε, μα ήδη έχουμε αρχίσει να το κάνουμε αυτό ιδιαίτερα με την ολοκλήρωση επιτυχών διαπραγματεύσεων με το ΑΕΜΟ και την ΚΑΟ. Του χρόνου όμως θα έχουμε ένα σημείο καμπής. Μετά από την επιστολή του κ. Γιούνκερ προθέσεων θα δώσουμε ξεκάθαρη πολιτική προτεραιότητα σε δύο θέματα που με αφορούν άμεσα σαν αρμοδιότητα. Το ευρωσήμα καταρχάς και μετά το ευρωπαϊκό διόδιο, το ευρωδιόδιο και η οδηγία του, ώστε να, να διευκολύνουμε την αρχή του χρήστης ή ο ρηπαίνων πληρώνων. Άλλες πρωτοβουλίες που θα αντιμετωπίσουμε το χρόνο ως τμήμα της, χαμηλής, της χαμηλών ρήπων είναι και αναθεώρηση της οδηγίας συνδυασμένων μεταφορών πρώτον, δεύτερον, νέοι κανόνες για την λειτουργία της αγοράς για λεωφορεία και επιβάτες και μετά βελτίωση και τα κίνητρα των δημοσίων, το διαγωνισμό του δημοσίου και των προμηθειών του. Το τρίτο ζήτημα που θα σας παρουσιάσουμε είναι πρωτοβουλίες για άλλες μάλλον πρωτοβουλίες για δικές μεταφορές. Επίσης, θα αντιμετωπίσουμε και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ως εξής θα αναθεωρήσουμε την ε, πρόσβαση όσον αφορά τα φορτηγά της ε, μεταφορές μακράς ε, απόστασης. Επίσης, άλλες δύο πρωτοβουλίες έχουμε για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Καταρχάς, η εκπαίδευση και τα προσόντα των οδηγών στις οδικές μεταφορές και μετά τα μέτρα για να βελτιώσουμε την ασφάλεια της οδικής υποδομής και των τούνελ των σειράγκων. Τώρα, θαλάσσιες μεταφορές. Του χρόνου είναι χρονιά της θάλασσας, οπότε θα έχουμε πολλές εκδηλώσεις, συναντήσεις, εργαστήρια, διασκέψεις. Οπότε θα ήθελα να δούμε την υιοθέτηση νέων πρωτοβουλειών όσον αφορά τους λίμενες υποδοχής, κατά προτίμηση το πρώτο τρίμηνο του 2017. Θα ελέγξουμε επίσης την υγεία και την κατάσταση της ε, θαλάσσιας νομοθεσίας και επίσης ανακοινώσαμε για το πρόγραμμα μας για το 2017 μια αναθεώρηση όσον αφορά τα σκάφη, τα μικρά σκάφη, τα επιβατικά. Ελπίζω πάντως τα οι επιτούτου εκδηλώσει κατά διάρκεια του έτου της θάλασσα να μα επιτρέψουν να εντοπίσουμε τα missing links στο θαλάσσιο τομέα, ώστε ακριβώ να ενσωματώσουμε πλήρω τον θαλάσσιο τομέα στο τομέα των πολυτροπικών υπηρεσιών και των πολυτροπικών λύσεων. Τώρα να περάσω στο επόμενο ζήτημα, στην αεροπλοεία. Η εφαρμογή της στρατηγικής για την αεροπλοεία θα μας απασχολήσει του χρόνου βέβαια διάφορε διαπραγματεύσει όσον αφορά τι αερομεταφορέ και την αεροασφάλεια και αντίστοιχε συμφωνίε με τρίτε χώρε θα είναι υπό εξέλιξη. Η Κομισιόν θα υθετήσει σύντομα την, πρόσταση, την πρότασή τη το 6 8 όσον αφορά τι αθεμητέ πρακτικέ και για το σιδηρόδρομο θα προτείνουμε επίση στο δεύτερο τρίμηνο του 2017 την αναθεώρηση του κανονισμού μας σε σχέση με τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρόμων. Καταλήγοντας λοιπόν, συγγνώμη λέει ο Επίτροπος, καταλήγοντας, όπως ακούσατε για το 2017 θα είμαστε έτσι αρκετά απασχολημένοι. Θα είναι πολύ σημαντικό για όλα τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα, Κομισιόν, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, να συνεργαστούν επικοδομητικά ώστε να διασφαλίσουμε τα σωστά παραδοτέα για το 2017. Βασίζομαι στην στενή σας συνεργασία και στην ενεργό υποστήριξη για να αποδείξουμε ότι η Ένωση μπορεί να κάνει διαφορά αν συνεργαστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε πάντοτε έτσι προς Θεού. Αλλά τέλο πάντων σας καλώ όλους να έχουμε ένα επικοδομητικό διάλογο με επιχειρήματα και έχοντας κατά νου συνέχεια ότι εμείς θέλουμε να πετύχουμε πράγματα στο τέλος. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ όλους σας και είμαι ανοιχτή για ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ε, παρουσίαση και για το γεγονός ότι ήσασταν ε, σύντομοι γιατί θα ακουστούν και διάφορα ερωτήματα. Να δώσουμε καταρχήν λοιπόν το λόγο στους συντονιστές, ξεκινώντας από Βίντου Βαντεκάβα. Ε, τρία λεπτά για τον κάθε ένα από τους συντονιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και την κυρία Πούλτσα ε, για τη σύντομη αλλά ξεκάθαρη παρουσίαση αυτή. Του χρόνου, εξ όσων καταλαβαίνω, θα έχουμε κάποια μεγάλα κομμάτια να επεξεργαστούμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό. Λίγο αισιόδοξη σας βλέπω όμως σε ό,τι αφορά τα αυτοκινούμενα οχήματα για το 17-18 στους ευρωπαϊκούς δρόμους, αλλά τι να κάνουμε, οι πολιτικοί χρειάζονται και αισιοδοξία. Κάθε επιτυχία λοιπόν σας εύχομαι. Σε ό,τι αφορά τώρα το πακέτο χαμηλών εκπομπών και τη σχετική τροπολογία, ελπίζω να μείνετε λίγο εντός χρονοδιαγράμματος. Γιατί οι πρωτοβουλίες, οι σε διάφορες περιστάσεις ε, προεξαγγέλλονται, αλλά διαρκώς αναβάλλονται στη συνέχεια. Από 1η Ιανουαρίου θα ξεκινήσει και το δεύτερο ήμιση της θετίας. Ελπίζω να μπορέσετε να τηρήσετε λοιπόν το αρχικό σχεδιασμό. Και σε θέματα εφαρμογή έχω μεγάλα ερωτηματικά και πολλέ υποσημειώσει, γιατί βλέπουμε ότι πολλά κράτη-μέλη υστερούν σε θέματα εφαρμογή. Και εδώ να είμαστε και ειλικρινεί και νομίζω ότι είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσει την ε, εφαρμογή. Τρία λεπτά έχω. δεν έχω άλλη ώρα τότε δηλαδή. Αλλά θα συνεχίσω λίγο. Μου λείπει το σκιάλο των επενδύσεων. Να είμαστε ειλικρινεί. Η διάδρομη TNT και το ΣΕΦ και το ΕΦΣΥ συνεπάγονται πολλέ θέσει απασχόληση και ο κόσμος περιμένει και κυρίως οι νέοι περιμένουν τις θέσεις απασχόλησης αυτές. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσετε να δίνετε προσοχή προς αυτά και μία ερώτηση να κάνω ειδικά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Κίνα. Ξέρω ότι δραστηριοποιείστε ιδιαιτέρως ε, υπέρ των σχέσεων αυτών με, τις, με την Κίνα. Αλλά και παραλλήλου μας ε, ανησυχούν οι επενδύσεις της Κίνας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη κυρίως και κυρίως σε ό,τι αφορά το fair play και σε ό,τι αφορά την ενιαία αγορά, οι Κινέζοι είναι πρόσδεκτοι. Αλλά στην ευρωπαϊκή συνδρομική βιομηχανία υπάρχουν ανησυχίες για το κατά πόσο είναι ισότιμη η όρια ανταγωνισμού. Πείτε μας λοιπόν. Και πάλι, επαναλαμβάνω ότι δεν μιλάω για προστατευτισμό Μιλάμε για την δίκαιη κατανομή τη αγοράς. Και κάτι άλλο, αν και δεν είναι στο χαρτοφυλακείο σας, τι γίνεται μεταξύ Boeing και Airbus. Αυτό παραμένει ένα σημείο ε, που επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Τα πράγματα αλλάζουν από μήνα σε μήνα και ενδεχομένω να διαμορφωθεί διαφορετική κατάσταση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε την καταγραφή του χρόνου. Κύριε Σέρτουκ, σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια και να θέσω τα ερωτήματά μου. Προτού μάλλον κοιτάξω ένα προς ένα τα θέματα, θα μου επιτρέψετε και θα κατανοήσετε να, ότι θα αναφερθώ σε αυτό που έγινε στη Γερμανία. Θα το αρνηθείτε βέβαια, αλλά ξέρω ότι η υπηρεσία σας δεν ήταν αναμεμειγμένη στη λήψη της σχετικής απόφασης, αλλά το λέω ξεκάθαρα ότι αυτά που έγιναν με τον ε, κύριο Γιούνκερ, με την ε, τηλέφωνο, με την ε, κυρία Μέρκελ και τον κύριο Τόπνεκνεκ, δεν συμβάλλουν στη διαφάνεια που είχε θέσει ως στόχο του τότε ο κύριος Γιούγκερ για να δώσουμε, να ενάψουμε και στον κόσμο να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό. Και δεν ήταν αυτό το οποίο προεξανήγγειλε στο πρόγραμμα του κύριος Γιούγκερ. Στο επόμενο θέμα, σε ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές, είπατε κυρία Επίτροπε, και θα ήθελα να μας πείτε για τα αυτοκινούμενα οχήματα Ίσως δεν το κατάλαβα, αλλά τι γίνεται. Τι προγραμματίζει συγκεκριμένα για το χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι ξέρετε ποιο είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχουμε για το θέμα αυτό. Το BM, η BNI για παράδειγμα, το 2017 είπε ότι θα χρησιμοποιήσει το Μόναχο ως πόλη για την διεξαγωγή δοκιμών. Αυτό κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση. Και για ένα άλλο θέμα να πω δύο λόγια. Να πάρω παράδειγμα την γερμανική πολιτική ηλεκτρονική κινητικότητα, ηλεκτρονική, ηλεκτρική συγγνώμη, κινητικότητα. Αυτό τι σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή τεχνολογία για τις μπαταρίες έχει μείνει πίσω και έχουμε κορυφαίους πολιτικούς ε, στη Γερμανία και υπουργό οικονομικών μεταξύ άλλων που καλεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία να προχωρήσει προς την έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή. Εσείς πώς το τοποθετήσετε γι' αυτό. Και να επανέλθω και στο θέμα των αεροπορικών μεταφορών αναφέρεται τους διάφορους κανονισμούς. Αλλά αυτό που εξακολουθεί να λείπει είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ξέρω τι προβλήματα αντιμετωπίζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Better Regulation, αλλά εδώ και 1,5 έτο ε, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι από εσά προσωπικά, να μα πούν τι θα γίνει. Αυτό το περιμένει και ο πολιτικό ο κόσμο, αλλά και ο οικονομικό κλάδο, Περιμένει να δραστηριοποιηθείτε για την 868, ε, τον 868 κανονισμό και για τον κανονισμό, για την ιδιοκτησία. Για τον 1088 είχαμε ακούσει κάτι πριν από δύο χρόνια, αλλά δεν έχουμε κάτι καινούργιο προς το παρόν. Τι θα γίνει, θα γίνει τίποτα στη θητεία αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσάκη Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ήρθατε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για το feedback. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε βέβαια τι θα μας υποβάλλετε λεπτομερέστερα ως προτάσεις για τη χρονιά της θάλασσας. Για τις μεταφορές είναι σημαντικό να δούμε ακριβώς πόσο σημαντικές είναι οι θαλάσσιες μεταφορές διεθνώ για μας και για όλους. Εμείς θα πρέπει να είμαστε σε θέση λοιπόν να προωθήσουμε τις θαλάσσιες μεταφορές σε όλη την Ένωση. Είναι ένα κρίσιμη σημασία τομέας για τα αυτοκιμένα οχήματα που αναφέρατε και τεχνολογία. Νομίζω εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικέ πτυχέ. Η μία πτυχή αφορά τι δημόσίε μεταφορέ. όπου βέβαια υπάρχουν διάφορε απόψει. σε σχέση ή σε αντίθεση με τι ιδιωτικέ μεταφορέ. Οπότε θα πρέπει εμεί να είμαστε ξεκάθαροι για ποιο είδο μεταφορών μιλάμε, για, τις, για τα γιοταχή, για τι δημόσιε μεταφορέ, γιατί ακριβώ. Οπότε και πάλι αναμένουμε περισσότερε πληροφορίε γι' αυτό. Τώρα κάποια άλλα πράγματα να προσθέσω. Σε σχέση με την ΙΚΑΟ, μας είπατε κάποια πράγματα τα οποία είναι ευπρόσδεκτα και είναι ένα από τα πιο θετικά που είχαμε φέτος. Παρ' όλα αυτά, λαμβάνουμε μεικτά μηνύματα όχι από εσά, από αλλού. Και ομολογώ ότι ενησυχώ όταν λαμβάνω μεικτά μηνύματα όταν δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και δεν έχουμε κάτι σαφές που καταλαβαίνουν και αποδέχονται όλοι. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει ε, μια ιδέα, μια αντίληψη ότι μπορεί να συνεχίσουμε με το παλιό EQTS, κάτι το οποίο δεν είναι στο θεματολόγιο μας. Γιατί νομίζω ότι οι μεταφορές τότε στο εσωτερικό της Ένωση θα μείνουν με μια μορφή που στην ουσία είναι απώλεια χρόνου και θα οδηγήσει σε θέματα ανταγωνισμού. Οπότε το θέτουμε αυτό σε εσά και είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι ήδη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Τώρα για το πακέτο των αερομεταφορών έχουμε καθυστερήσει στη ψηφοφορία για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι ο συγητής έκανε θαυμάσια δουλειά εδώ. Έκανε πολύ καλή δουλειά και την αποδεχόμαστε οι περισσότεροι. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις κοινέ αρμοδιότητε με άλλε επιτροπές, όχι με την άποψη των γνωμοδοτήσεων α πούμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μην έχουμε μόνο με τον πρόεδρο της Επιτροπής, αλλά όλη την Επιτροπή και να δούμε ακριβώς τι επιρροή θα έχει η Επιτροπή με την πραγματογνωμοσύνη σε συγκεκριμένους τομείς και αν γίνεται στους περισσότερους. Τώρα το άλλο που αναφέρατε για την, για την αρμοδιότητα, νομίζω στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να δική μας αρμοδιότητα, παρά τις παρόν τρεις επιτροπέ να συμμετέχουν και αυτές το ΙΣΕΡ επίση για όλα αυτά που θα γίνουν του χρόνου σα ευχαριστεί και θα περιμένουμε για του χρόνου ακόμα περισσότερε πληροφορίε από εσά. Ευχαριστώ πολύ. Η το λόγο. Ε, ευχαριστούμε ε, κύριε Επίτροπη και από την πλευρά των ε, φιλελευθερών για την παρουσίασή σας. Να θέσω και εγώ τα δικά μας ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική CITS. Ναι, γνωρίζουμε όλοι μας ότι αυτό είναι το μέλλον, δηλαδή να έχουμε συνδεδεμένα αυτοκίνητα τα οποία εν μέρει είναι αυτοκινούμενα, αυτοοδηγούμενα, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχετε δεσμεύσει, αν θέλετε, το κατάλληλο εργατικό, αν θέλετε, δυναμικό, ε, νομικού δηλαδή, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τα ζητήματα, για παράδειγμα, τη ασφάλιση. Ποιο θα έχει την ευθύνη, για παράδειγμα, σε περίπτωση ατυχήματο σε ό,τι αφορά αυτά τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα. Άρα, λοιπόν, το ερώτημα που ε, θέτω είναι, έχετε ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα, με αυτέ τι πτυχέ. Δεύτερο ε, θέμα τώρα είναι τα διόδια και αναφερθήκατε σε αυτό, δηλαδή πάντοτε ο στόχο σα ήταν να ακολουθήσουμε την αρχή ορυπαίνων πληρών και αυτό είναι και ο δικός μας στόχος, δηλαδή να μπορέσουμε να να, να μπορέσει να συμμερφωθεί η αγορά με αυτόν τον με αυτή την αρχή. Αλλά η συμφωνία η οποία τελικά συνάφθηκε ε, ε, και μάλιστα δύο φορές ε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έτσι κάπως σκοτεινά, δεν μας άρεσε και εμάς και θα πρέπει δηλαδή να ελεγχθεί και από εσά από την αρμόδια επίτροπο κατά πόσο μια τέτοια συμφωνία είναι νόμιμη καλό θα ήταν πάντως να σχολιάσετε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή έγινε μια διαπραγμάτευση από, το, από την πλευρά της ε, Επιτροπής και από το δικό μας ε, Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Στομπλέντα, από την πλευρά της Γερμανίας, χωρίς να λάβει ε, χώρα μια συζήτηση εδώ χωρίς να υπάρξει και σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, κάποια ακόμα σημεία. Το ECMR, δηλαδή τα ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικές φορτωτικές ή μεταφορικά έγγραφα αυτό ε, ξεκίνησε ε, σε επίπεδο, ως πρωτοβουλία δηλαδή, σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, αλλά θα έπρεπε να ε, χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε εσωτερικές μεταφορές, εμπορευματικές μεταφορές ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε ξεκινήσει κάποια προσπάθεια εδώ, ε, για παράδειγμα, να απευθυνθείτε στις χώρες οι οποίες δεν έχουν κυρώσει την κατάλληλη, τη σχετική συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών. Και από εκεί και μετά υπάρχει και μια σχετική συμφωνία σε ό,τι αφορά τους λιμένες, την οποία δεν έχουν κυρώσει μια σειρά από κράτη-μέλη. Μας είπατε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως θα δώσει προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα αλλά δεν θα πρέπει να ξεκινήσει η Επιτροπή να αποστέλει αυτές τις επωνομαζόμενες εμπλέ επιστολές στα κράτη-μέλη που δεν έχουν ανταποκριθεί σχετικές τους υποχρεώσεις ε, κύρωσης. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό 868 και το ναυτιλιακό έτος ε, μετά δηλαδή από το ε, πακέτο για τις ειδικές μεταφορές, πότε θα έρθουν, αυτό αναμένουμε όλοι μας. Και σε ό,τι αφορά το ΣΕΣ του ΠΛΑΣ και τα, την οδηγία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών ε, στην αεροπορία, ποια είναι η συνέχεια που θα δοθεί σε αυτούς τους τομείς. Ίσως, ε, για παράδειγμα, με τη νέα Ισπανική κυβέρνηση είπατε ότι έχει υποθεί από κάποιους ότι ενδεχομένω να υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει πάλι να δοθεί όθηση στις διαπραγματεύσεις. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε κάτι κι εσείς από την πλευρά σας. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Επίτροπε. Χαίρομαι που τώρα το καμποτάζ, το καμποτάζ ήταν, είναι μάλλον ψηλά στην ατζέντα, στο θεματολόγιο. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι η υπόθεση αυτή αφορά πολλές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν αθέμητο ανταγωνισμό λόγω ακριβώς έλλειψης Νομοθεσία στον τομέα του καμποτάζ. Σήμερα έχουμε και κοινωνικό dumping και υπάρχει νομοθεσία που επιτρέπει δυστυχώ τη διαιώνιση αυτή τη κατάσταση, η οποία είναι πολύ άσχημη. Εγώ ήμουν μεταφορέας, έκανα διεθνεί ε, μεταφορέ. και νομίζω ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το παρελθόν και έχει φτάσει σε μια σχεδόν εγκληματικά. Δηλαδή η κατάσταση αυτή σκοτώνει στην ουσία, εξοντώνει τις εταιρείε οδικών, διεθνών οδικών μεταφορών. Οπότε, ερώτησή μου, πότε θα μας υποβάλλετε τις προτάσεις σας συγκεκριμένα για το καποτάζ και βεβαίως ε, πότε θα μας υποβάλλετε το γενικότερο πακέτο για τις οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Ε, τώρα, επόμενοι ομιλητές, 1,5 λεπτό έχουν στη διάθεση ναι, θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα να συμφωνήσω με του δύο Γερμανού συναδέλφου που πριν από μένα το λόγο και αναφέρθηκα στο ζήτημα των γερμανικών διοδίων. Ε, παρότι λοιπόν τα άτομα τα οποία θύχτηκαν ε, σε σχέση με αυτή τη διαπραγμάτευση ανήκουν ε, στη δική μας πολιτική ομάδα, θα πρέπει να πω ότι μετά από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν και σε επίπεδο της, του Ευρωπαϊκού Σώματος Κυκλοφορίας της Eurovignette, ότι είμαστε λίγο σκεπτικοί, γιατί πραγματικά θα πρέπει αυτή η πρωτοβουλία να αποτελέσει τον ακρογωνίο λίθο της προσπάθειας που κάνουμε. Δεν αντιλαμβανόμαι λοιπόν το πώ κινήθηκε σε αυτό το επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτή μια τέτοια προσέγγιση. Από εκεί και μετά Ε, με βάση τη νέα ε, συμφωνία ουσιαστικά ε, οι χρήστες των οδικών δικτύων στη Γερμανία όχι μόνο θα τα βάλουν τα σχετικά διόδια, ενδεχομένω να πιστωθούν και με αυτά. πράγματα το οποίο βέβαια δεν ευθυγραμμίζεται καθόλου και με τις πολιτικές μας σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει πλήρης αδιαφορία. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι ως Γερμανός αυτοκινηστής θα πρέπει να λαμβάνω ε, μια τέτοια επιστροφή σε επίπεδο ιδιωτήτων μόνο και μόνο λόγω της εθνικότητάς μου ε, ε, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορεί να, να, είναι κάτι τέτοιο δίκαιο. Είναι, δεν είναι σε καμία περίπτωση ικανοποιητικό κάτι τέτοιο. Αυτά πολύ σύντομα να κάνω όμως και ένα θετικό σχόλιο να σας ε, ε, συγχαρώ ε, ε, ω προ τι προσπάθειε που κάνετε στο επίπεδο των εκπομπών και του λαμβάνετε υπόψη τι δικέ μας ε, απόψει. και επίση θα θέλαμε να ακούσουμε σε σχέση με τα μία επαντρωμένα αεροσκόπητα drones, τι συμβαίνει σε δικό σα επίπεδο και με το Συμβούλιο και θα θέλαμε να μας κρατάτε ενήμερο σε σχέση με αυτέ. τις συζητήσει. Γεια σας κύριε Επίτροπε, χαιρόμαστε που σας βλέπαμε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Δύο σύντομε ερωτήσει για θέματα οδικών μεταφορών. Καταρχά, Είδαμε ενδιαφέρον την πρόσφατη έκθεση και την έρευνα της Κομισιόν σε σχέση με τα δεδομένα που αφορούν τις συγκρούσεις και τα, και τα ατυχήματα, σοβαρές ε, βλάβες, τραυματισμούς κτλ. Έχετε στοιχεία πέραν από τα θύματα όσον αφορά τους σοβαρούς τραυματισμούς. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε συχνά και με τις αστικές περιοχές και τώρα το χειμώνα κινδυνεύουν ιδιαίτερα και οι τα παιδιά κτλ. Και, και για το Uber θα ήθελα κάποιο σχόλιο σε σχέση με την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπου συζητήθηκε το κατά πόσο είναι μόνο η ηλεκτρονική πλατφόρμα ή η υπηρεσία μεταφορών του Uber. Βέβαια, εμεί στην Ιρλανδία θεωρούμε το εκτό απολαθούμε ηλεκτρονική είναι και η υπηρεσία μεταφορών. Οπότε θα πρέπει να υπάγεται και να υπόκειται σε όλη την νομοθεσία για του κανονισμού για αυτό το τομέα στι διάφορε χώρε. Επικτείνονται ταχύτητα στην χώρα μου και συχνά έχουν οδηγού που δουλεύουν πάρα πολλέ ε, ώρε και δεν βγάζουν πολλά χρήματα. Θα ήθελα λοιπόν να τα σχολιάσετε όλα αυτά. Επίση, να μα πείτε κάτι για την έρευνα που αφορά αυτό που είχαμε πει ότι στο τέλο 15 θα γίνει για περισσότερη εξέταση του θέματο του Uber. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο καταρχά και την συγχαίρω για τη δουλειά τη. Για τα συνδεδεμένα οχήματα, τα αυτοματοποιημένα, το 17 είναι σημαντική ημερομηνία. Και επίση για το πακέτο θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αλλά δεν υπάρχει μετάφραση στα αγγλικά, λέει η Επίτροπο. Ε, δεν ακούω καλά. Μόνο ένα έτσι μακρινό θρόισμα. Α, τώρα, τώρα κάτι ακούω, κάτι ακούω. Να τα ξαναπώ, λέει ο πρόεδρος στα γερμανικά. Μάλλον ο μιλής στα γερμανικά. Κρίμα, κρίμα που δεν ακούσατε. Γιατί ξεκίνησα ακριβώ με τα συγχαρήκια. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνατε λοιπόν. Και ξαναλέγα, ξαναλέω, το 17 είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι κοντά. Και συγχαρητήρια για τις ε, προσπάθειές σας για, αυτή, για τον τομέα των οδικών, για το πακέτο απαραίτητα, για όλο τον τομέα των οδικών μεταφορών. Επενδύσεις τώρα στις υποδομές. Στα πλαίσια λοιπόν της λογικής εργασίας θα πρέπει να προβλέψουμε τι γίνεται με το επόμενο πολιετές χρηματοοικονομικό πλαίσιο και τα μελλοντικά εργαλεία, τα οικονομικά. Εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα του ευρωσήματος. Συνεργατική οικονομία. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσετε και θα πρέπει να λάβετε μια κανονιστική θέση για αυτό το θέμα, γιατί βλέπουμε ότι απασχολεί πολύ όλες τις χώρες μέλη. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η συνεργατική οικονομία στηρίζεται πάρα πολύ στις μεταφορές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει τουλάχιστον μια οδηγία για αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι η οικονομία χρειάζεται ε, υπηρεσίες προς πολίτες παντού σε όλες τις χώρες. Τι θα λέει ε, κύριε Επίτροπε, η δική μου ερώτηση έχει να κάνει με αυτήν που έθεσε η Λούση Άντερσον. Δηλαδή, υπήρξε η δημοσίευση μια ε, μελέτη σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ατυχημάτων ε, του συμπτώνου και γίνονται κάποιε προτάσει για τη μείωση, ειδικότερα των σοβαρών ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, γίνεται εκεί μια ε, αναφορά σε ό,τι αφορά και τον στόχο που θα πρέπει να θέσουμε σε ό,τι αφορά δηλαδή τη μείωση των σοβαρών των ατυχημάτων και τώρα θέλουμε να υπάρξει ένας νέος στόχος σε ό,τι αφορά τα σοβαρά ατυχήματα. Οπότε πότε να αναμένουμε μια τέτοια πρόταση από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά δηλαδή τη μείωση των σοβαρά τραυματισμένων. Και εδώ σας υπενθυμίζω και την πρόταση που είχαμε κάνει το 2011 όπου προβλεπόταν δηλαδή να στόχο στη τάξη του 40%. Ευχαριστώ biztos asszony. Ευχαριστούμε και εμείς. Szeretnék kettő mondatot szólni, amit... Θα ήθελα και εγώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο ε, και ειδικότερα σε σχέση με ένα ζήτημα το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένα στο, στο παρελθόν ένα ε, είδος ε, συνδρομής ε, σε έναν ευρωπαϊκό χάρτη το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνδρομικές μεταφορές ε, αλλά και σε άλλες. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο ε, να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα ενό ε, ειδικού εισιτηρίου, για παράδειγμα στου ε, νέου μα, ούτω ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. οι συνάδελφοι εδώ που συμμετέχουν στην Επιτροπή Τραν γνωρίζουν αυτή την πρόταση. Και παρότι γνωρίζουμε ότι δεν είστε η μόνη αρμόδια επίτροπος για το λόγο πρόγραμμα, έχετε πραγματικά δείξει πολύ θετική στάση, το έχετε υποστηρίξει ε, στο παρελθόν και γι' αυτό θα θέλαμε να μας πείτε αν θέλετε να κάνετε κάτι σε σχέση μας στο, στο μέλλον. Ο κύριος ε, Γιούγκερ είχε αναφερθεί άλλωστε και εκείνος από την πλευρά του σε αυτό το ζήτημα. Εγώ δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσω γιατί πρέπει να πάω σε άλλη συνεδρίαση, αλλά χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα μαζί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε για το πρόγραμμα εργασία για του χρόνου, όπως η Λούση, να ρωτήσω τι γίνεται με τα σοβαρά ατυχήματα και του, τραυματισμούς, σοβαρούς τραυματισμού, γιατί μιλήσατε για το θέμα των συνδεμένων των αυτοματοποιημένων αυτοκινήτων και η χρήση τη τεχνολογίας για τη μείωση δηλαδή των ατυχημάτων και των θανάτων με αυτόνομα συστήματα πέδηση ταχύτητας, κλπ. Να μας πείτε ακριβώ πώς προσδιοθέστε να προχωρήσετε εδώ σε αυτό το τομέα μαζί με αυτό το πακέτο ασφάλειας, το safety package. Για την αεροπλοεία κάναμε πολλές συζητήσεις και ανταποκριθήκαμε βέβαια στην σταρική σας η οποία είναι ευπρόσδεκτη. Θα αναθεωρηθεί βέβαια κάποια στιγμή του χρόνου και θα είναι καλό αυτό. Βέβαια το θέμα είναι τι γίνεται με τα άλλα πακέτα, SS2, τα σλότς, τι μπορεί να γίνει με αυτά. Και να σας ευχαριστήσω που απαντήσατε στην προφορική ερώτηση στο Στρασβούργο πριν εβδομάδες και να γνωρίσατε την ανάγκη ενημέρωσης των μελών του Κοινοβουλίου για αυτές τις διαπραγματεύσεις που δεξάγονται. Και ξέρουμε ότι ό,τι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή εκτός ενώσης στο των της είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ο κύριο Φαμιλτμπέργκ. Στα Ολλανδικά. Και εγώ ανησυχώ για τη συμφωνία που έγινε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπή και Γερμανίας για τα γερμανικά σχέδια για τα διόδια. Πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται. Υπάρχουν ε, στοιχεία που συμβάλλουν στην διακριτική μεταχείριση των χρηστών των δρόμων μας και γιατί πιστεύετε ότι το γερμανικό σχέδιο δεν θα υπονομεύσει τη δική σα στρατηγική για τι χαμηλέ εκπομπέ. εκπομπές. Εγώ αμφιβάλλω ιδιαίτερο τρίτο σημείο. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, μεταξύ άλλων και η Ολλανδία, αλλά και η Αυστρία και άλλε χώρε που έχουν ανακοινώσει ότι θα προβούν σε νομικέ ε, ε, ενέργειε. Ξέρω ότι έχετε νομική υπηρεσία και έχετε λάβει νομικές γνωμοδοτήσεις. Πείτε μας λοιπόν πώς ε, αξιολογείτε τις χώρες αυτές που θέλουν να υποβάλουν ένσταση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και ένα άλλο θέμα το οποίο το έθιξε και η κυρία Μέιζερ, η συνάδελφο, το Single European Sky 2 Plus και τα δικαιώματα των επιβατών. Έχουμε πάρα πολλά μεγάλα πακέτα τα οποία έχουν παραλύσει στην παρούσα φάση στο Συμβούλιο. Μήπως δεν έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να ξεκινήσετε εσείς ένα σχέδιο δράσης. Δύο στοιχεία θα πρέπει να λεφθούν υπόψη, θεωρώ το θέμα του Γιβραλτάρ, το οποίο θα πρέπει να προσθεθεί στο, ε, στην ατζέντα του Συμβουλίου, το γενικότερο θέμα του ενέργειου χώρου, αυτό θα γλιτώσει ε, και πάρα πολλά χρήματα, αλλά και πάρα πολλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Και μήπως θα πρέπει σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο να διοριστεί ένας ειδικός εντεταλμένος για να διαμεσολαβήσει σε ό,τι αφορά τον αέριο χώρο του Γιβραλτάρ και να βρεθεί μια λύση, γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεπρέης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπούλτς και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι έρχεστε συχνά στην Επιτροπή μας και αυτό πραγματικά ευνοεί την επικοινωνία. Να τονίσω το θέμα του βασικού κανονισμού της ΕΑΖΑ. Εσείς ε, αναφερθήκατε στα θέματα του δικαίου ανταγωνισμού και ο συνάδελφο Έρτουγκ μίλησε για το σχετικό κανονισμό των 10.08. Θα ήθελα να σας πω ότι στην Επιτροπή αποφασίσαμε μια κανονική διαδικασία να ακολουθηθεί για την ΕΑΖΑ, όχι μόνο από τη δική μου ομάδα, αλλά και από τις άλλες ομάδες σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Σας παρακαλώ λοιπόν να το λάβετε η υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενο μελητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Επίτροπε, για τι εξηγήσει αυτέ. Για τι γερμανικά διόδια, νομίζω είπαν οι συνάδελφοι αυτά που τα να υποθούν. Οι γειτονικέ περιοχέ ε, και οι γειτονικέ χώρε τη Γερμανία ε, έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Και νομίζω ότι θα πρέπει να η δράση. Δύο ερωτήσει. Καταρχά ε, για τα θέματα των, των δικαιωμάτων των επιβατών. για την ε, κατάρτιση των δικαιωμάτων ε, των συνδρομικών ε, επιβατών. Μια και το Γερολιτάν δεν συνδέεται με συνδρόμου, ελπίζω να προχωρήσουμε εδώ. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι στους διάφορους τρόπους μεταφορών. Υπάρχει το θέμα των αποζημίωσεων και το καθεξής εδώ πέρα. Πώς σκέφτεστε να επιβάλλετε ίσους όρους ανταγωνισμού. Και δεύτερη ερώτηση. Πριν από 8-9 ε, μήνες ως Κοινοβούλιο καταρτήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για το θέμα της, των συνδρομικών μεταφορών. Και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τις ε, επενδύσεις από την Κίνα. Και τώρα λοιπόν υπάρχει κίνδυνος ο εξή να μην σημειωθεί πρόοδος, να μην ξέρουμε πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Εσείς ως Επίτροπος ε, για θέματα μεταφορών ε, είσαστε αναμειγμένοι σε τέτοια θέματα σε ό,τι αφορά την επαναβιομηχανοποίηση σε θέματα. Συντρεζόμουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γιούτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ είμαι εδώ με Επίτροπο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες στον τομέα της αεροπλοείας. Υποφελούμε σε για να επαναλάβω κάποιες αρχές που σας ανέφερα και πριν δύο εβδομάδες στο Στρασβούργο. Αρχές που μας είναι προσφυλής. Κοινωνικά δικαιώματα και αθεμητός ανταγωνισμός. Και μάλιστα πρόσφατα διαβάσαμε στον τύπο στην Ιταλία ότι η Etihad θα μπορούσε στην Ιταλία να απολύσει 2.000 προσωπικό για εξυγένση. Εταιρεία που έχει κονδύλια από τρίτες ε, χώρες και που έχει αγοράσει την Αλιτάλια μετά από βούληση της ε, Ιταλικής κυβέρνησης και επικύρωση της Κομισιόν που έδωσε θετική γνώμη για την αγορά αυτή. Παραχωρούμε λοιπόν όλο και περισσότερο έλεγχο της αγοράς μας και μετά απολύουμε 2.000 κόσμο. Αναρωτιέμαι λοιπόν εγώ, με ποιο τρόπο προτίθεστε να προστατεύσετε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης ενώπιον κεφαλαίων τρίτων χωρών που δεν υπόκεινται στους ίδιους κανόνες για, για κρατικές ενισχύσεις που πρέπει να τηρήσουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πώς θα αποφύγουμε την εξάρθρωση των επιχειρήσεών μας και πώς θα διατηρήσουμε την δουλειά των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορούμε να αναμένουμε συγκεκριμένα μέτρα εκ μέρους της Κομισιόν για αυτό το θέμα, πέραν των διμερών συμφωνιών, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εγώ χαίρομαι για την παρουσία σας σήμερα και είμαι σίγουρος πως το παράπονο ότι μόνο έξι φορές μας είδατε θα φροντίσει ο Πρόεδρος να τις κάνει περισσότερες τον επόμενο χρόνο. Θα αναφερθώ και εγώ στην αναθεώρηση του κανονισμού 1072 για τις διεθνείς οδικές μεταφορές. Ξέρουμε ότι κάποιες ε, διατάξεις των ενδομεταφορών αυτών ε, δεν μπορούν να ελεγχθούν από τους μηχανισμούς των κρατών μελών, είτε διότι κάποια στοιχεία είναι εύκολα να παραποιηθούν, είτε η γενική αδυναμία αυτών των ελέγχων. Αυτό έχει οδηγήσει κάποια κράτη-μέλη σε έναν ιδιότυπο νέο προστατευτισμό. Κάθε κράτος παίρνει μονομερός κάποια μέτρα, τα οποία επιδρούν όμως στα αλλοδαπά οχήματα. Παίρνοντα σαν δεδομένο την δυσκολία των μηχανισμών ελέγχου, μήπω οι κανονισμοί μα θα έπρεπε να εμπεριέχουν αυτή τη δυσκολία και να πηγαίνουν ακόμα παραπέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε στη σημερινή μα ε, συνεδρία. Έχω ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά το πακέτο για τι οδικέ μεταφορέ. Ε, γιατί προφανώ ε, υπάρχει και μια σημαντική κοινωνική διάσταση σε ό,τι αφορά ειδικότερα την οδηγία για του απασχολημένου εργαζόμενου. Και αφορά βέβαια και του οδηγού των λεωφορείων και το ελάχιστο εισόδημά του. Όπω θα γνωρίζετε, κύριε Επίτροπε, υπάρχει μια διαδικασία κατά παράβαση η οποία έχει ξεκινήσει σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Και το ερώτημά μου είναι το εξή. Θεωρείτε πω θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μια επιβράνδυση των διαπραγματεύσεων ή θα επιτευχθεί τελικά μια συμφωνία ε, ε, σε ό,τι αφορά το παλιό των οδικών μεταφορών, ε, αφού δεν έχουμε ακόμα λάβει μια οριστική απόφαση από την πλευρά του δικαστηρίου. Κύριε Ντεμόντι, ευχαριστώ πρόεδρε που ήρθατε. Επίτροπε που ήρθατε. Πολλά θέματα αναφέρθηκαν από του συναδέλφου και ενα αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ενέργειο χώρο. Τι γίνεται και τι κάνει η Κομισιόν εδώ. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια πρόσκληση στα πλαίσια της για την αεροπλοεία. Θα ήταν όμως καλό το συγκεκριμένο ζήτημα αυτό να έχει ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Μετά, να πω κάτι άλλο για την Κίνα και τις επενδύσεις της αλλά τα logistics, η επιμελητία αποτελούν και αυτό ένα τρόπο ελέγχου των συναλλαγών. Έχετε λοιπόν κάποια μελέτη αντικτύπου για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν και παραβιάσεις κοινωνικών δικαιωμάτων στα πλαίσια αυτών των συναλλαγών. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίασή σας, να θέσω και κάτα, κάποια ερωτήματα. Έχουμε αυτές τις επιχειρήσει ό,τι αφορά το λεωφορείο, το οποίο ζήτημα θα μπορούσαμε να λύσουμε με ταχογράφου και στα παλαιότερα και στα νέα οχήματα, έτσι ώστε να αποφύγουμε ότι ένα Ρουμάνος, για παράδειγμα, οδηγός λεωφορείου, να μετακινείται για παράδειγμα όλη την ώρα να οδηγεί στη Γερμανία και στις κάτω χώρες αλλά πληρώνεται με μισθου ε, Ρουμανίας. Ε, όπως για παράδειγμα και στη Ryanair το βλέπουμε δηλαδή ότι το 1 τρίτο των ε, πιλότων ουσιαστικά εργάζονται για άλλη επιχείρηση και ε, πληρώνονται ε, μόνο όταν πραγματικά πετούν. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγοί καλούνται να σκεφτούν το αν θα εργαστούν κάθε φορά για να δουν αν θα καλύψουν τα έξοδα τους ή όχι. Από εκεί και μετά ένα δεύτερο ζήτημα αφορά ε, τα διόδια και υπήρξε και ένα πολύ καλό άρθρο στην site της τελευταίας Κυριακής. Δηλαδή, αν ακολουθήσει, έλεγε το άρθρο, κάθε ε, χώρα ε, αυτήν την στατηγική, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, τη διακριτική μεταχείριση των υπηκών τη κάθε χώρα Δηλαδή, αν πήγουν τα αυστριακά πανεπιστήμια, εμεί θα χρεώνουμε όλου του ξένου φοιτητέ χιλιά ευρώ για δίδακτρα, αλλά του υπόλοιπου όχι, ή στα νοσοκομεία γίνει κάτι αντίστοιχο, τότε πραγματικά θα περιπλακούν τα πράγματα. Και όμω αυτό συνέβη στα διόδια. Δηλαδή, ουσιαστικά ε, ε, επιβαρύνονται άλλοι υπήκο περισσότερο σε σχέση με άλλου. Και αν, δεν, αν έχουμε μια τέτοια παραβίαση αυτή τη αρχή, αν δηλαδή υπερισχύσει ο εθνικό εγωισμό, πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση διαλυθεί. Γι' αυτό το λόγο δεν αντιλαμβάνομαι γιατί προέδρει αυτή την κίνηση ο πρόεδρος Γιούγκερ. Ε, γιατί πάντοτε προσπαθούσε να είναι αμερόληπτος και να μην προβαίνει σε διακρίσεις. και ε, πραγματικά ε, ε, ο κάθε ένας τώρα που δεν είναι Γερμανός μπορεί πράγματι να κάνει παράπονα σε ό,τι αφορά την καταβολή διοδίων στη Γερμανία. Οπότε θα ήθελα να μας, να μας να μας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε γιατί ε, πραγματικά δεν θεωρώ και δίκαια τη μεταχείριση τη δική σας ε, γιατί η απόφαση λήφθηκε από άλλους και καλείτε εσείς να αντιμετωπίσετε τώρα το τι συμβαίνει. Ε, πάντως σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί αυτό θα μας φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και δεν αποτελεί πρόοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί βήμα προς τα πίσω. Ακούσατε πάρα πολλά ερωτήματα κύριε Επίτροπε. Ο λόγος λοιπόν τώρα σας στάζει για να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Ε, κάθε φορά ε, νιώθω σαν να περνάω καινούργια ακρόαση όταν έρχομαι τη συμμετέχω σε μια συνεδρίαση εδώ Επιτροπή ε, του Κοινοβουλίου. Πάντω, θα προ... κάνω ό,τι καλύτερο για να απαντήσω στα ερωτήματα που θέσατε όσο γίνεται πιο διεξοδικά. Ναι, λέω πρώτο, αλλά ακρόαση ήταν εξαιρετική ούτω ή Ναι, τέθηκαν κάποια ερωτήματα σε ό,τι αφορά ε, τα αυτόνομα, ε, αυτοκινούμενα οχήματα. Οπότε. Ε, Αγαπητέ ε, ήθελα να σας πω ότι πραγματικά δεν είμαι τόσο φιλοδοξό, αν ενδεχομένω να ακούστηκα. Είπα απλώς ότι το νέο CITS αναφέρει μία ε, σειρά από υπηρεσίες οι οποίες θα οδηγήσουν στο πρώτο επίπεδο αυτοματοποίησης. Αυτό το πρώτο επίπεδο αυτοματοποίησης είναι τα διασυνδεδεμένα οχήματα. Σε αυτήν λοιπόν τη στρατηγική CITS απαριθμούμε όλες τις υπηρεσίες και όλες τις λειτουργίες οι οποίες καλύπτουν τα ζητήματα ασφάλειας, επιβολή δηλαδή της νομοθεσίας σε σχέση με ζητήματα ασφαλείας στον κώδικα οδική κυκλοφορία και μιλάμε για στοιχεία τα οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε ω το 2019. Το επόμενο βήμα από εκεί και μετά ε, αφορά τα συνεργαζόμενα οχήματα, cooperative Δηλαδή θα υπάρχει πλέον επικοινωνία μεταξύ τη υποδομή και του ε, οχήματο. Και η φιλοδοξία μας είναι ως το 2030 να ε, ολοκληρωθεί και αυτό το δεύτερο βήμα. Και από εκεί μόνο και μετά, δηλαδή στο τρίτο βήμα, περνάμε πλέον πραγματικά στην αυτόνομη οδήγηση των οχημάτων και εκεί τίθενται όλα αυτά τα ζητήματα νομικής φύσης και άλλα που αναφέρονται τόσοι από εσά. Ε, και εδώ πραγματικά δεν είμαι τόσο ε, φιλοδοξή. Δηλαδή ε, πλήρη αυτόνομη οδήγηση με όλα τα προβλήματα να έχουν επιληθεί αναμένω για το 2050. Οπότε πραγματικά το βάθος χρόνου είναι μεγάλο. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά τεράστια βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε. Και μην σκεφτείτε μόνο τη Γερμανία, σκεφτείτε τη Ρουμανία, σκεφτείτε τη Βουλγαρία, σκεφτείτε την Ελλάδα ε, και σκεφτείτε και όλες τις ε, χώρες συνοχής που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, για αυτό το πλαίσιο. Οπότε πραγματικά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Ε, το βαθμό απορρόφηση, αν θέλετε, αυτών των νέων τεχνολογιών δεν θα είναι ίδιο σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε, πραγματικά, όταν ε, αναφέρομαι σε μελλοντικό σχεδιασμό, αναφέρομαι ε, στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω ενιαίο χώρο μεταφορών. Αλλά από εκεί και μετά, βέβαια, κάποιε χώρε θα εφαρμόσουν πολύ ταχύτερα τα σχετικά συστήματα, γιατί θα είναι ε, έτοιμε νωρίτερα από ό,τι άλλε. Ε, για παράδειγμα, βλέπουμε να υπάρχει αυτόνομη οδήγηση σε πολύ ελεγχόμενε ε, περιοχέ, για παράδειγμα σε αεροδρόμια, σε πανεπιστημιακά κάμπου. Αλλά η προσέγγιση μα θα είναι σταδιακή. Τώρα, σε ό,τι αφορά δημόσια έναντι ιδιωτικής πρωτοβουλία. Ε, και βλέπουμε εδώ πραγματικά μια σειρά από πρωτοβουλίε οι οποίε ε, προκύπτουν όχι μόνο σε ό,τι αφορά νέων λειτουργιών ε, των οχημάτων, αλλά και σε συνέχεια των ψηφιακών πλατφορμών. Δηλαδή υπάρχουν πολλά περισσότερα πλέον συμμετοχικά μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται ειδικότερα σε πόλει και είμαστε υπέρ αυτών των μοντέλων χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αυτά τα μοντέλα προωθούν την ε, συνδεδεμένη, την αυτόνομη οδήγηση. Απλώς βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και της ε, χρήσης των αυτοκινήτων. Και βλέπουμε αυτά τα συστήματα να εφαρμόζονται και οι λύσεις ε, στις πρωτεύουσε και βλέπουμε να καθίστανται όλο και περισσότερο ε, ηλεκτρικά τα οχήματα. Και βέβαια και αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική μεταβολή την οποία προωθούμε και η οποία βλέπουμε να συντελείται, δηλαδή μετάβαση προς οχήματα μηδενικών εκπομπών, ε, δηλαδή ηλεκτρικά κινούμενα οχήματα. Και εδώ αναφέρομαι πάντως στις οδικές μεταφορές. Ε, δηλαδή σε ό,τι αφορά την αεροπορία έχουμε να κάνουμε κυρίως με βιοκαύσιμα και σε ό,τι αφορά την αυσυπλοεία έχουμε να κάνουμε κυρίως με εγκροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG. Επιτρέψτε με τώρα να περάσω σε ένα άλλο σχετικό με αυτό ζήτημα του electrification, δηλαδή της ε, μετάβασης στην ηλεκτρική ενέργεια. Προφανώς ε, ε, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους και στις δημόσιες μεταφορές να προωθήσουν αυτό την, την μείωση δηλαδή της, των εκπομπών άνθρακα και την 1η Δεκεμβρίου είχαμε την παρουσίαση ενός νέου εργαλείου για την χρηματοδότηση των νέων καθαρών οχημάτων την 1η λοιπόν Δεκεμβρίου μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Transport Council κάναμε αυτή την ανακοίνωση και ήδη έχουμε τρεις πολύ καλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν τύχη και έγκρισης. Μία από αυτές μάλιστα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Ε, για την παροχή ακριβώς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο δηλαδή των οδικών ε, μεταφορών. Για παράδειγμα στη Ρήγα υπάρχει ακριβώς ε, μια τέτοια υποδομή που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την κίνηση οχημάτων. Υπάρχουν και αντίστοιχα οχήματα που έχουν ξεκινήσει στη Γαλλία και στην Ισπανία και ενθαρρύνουμε τις πόλεις να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να κάνουν συλλογικές παραγγελίες της σχετικής υποδομής ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερες τιμές από την ε, βιομηχανία. Άρα λοιπόν βλέπουμε να κινούνται εδώ τα πράγματα στι ε, πόλει, αυτό μας ενθαρρύνει και θα, είμαστε, θα στοχεύσουμε τι προσπάθειές μας ώστε να καλύψουμε τα κοινά που θα προκύψουν σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των δημοσίων μεταφορών, έτσι ώστε να επιτύχουμε αποτελεσματικότερη ψηφιοποίηση και μείωση των κομπών άνθρακα στι μεταφορέ όπω είχαμε ανακοινώσει στην πολιτική μα. Τώρα, επιτρέψτε με να περάσω στην ε, περίπτωση τη Boeing και τη Airbus ε, δύο δηλαδή προετοιμαζόμενες ε, περιπτώσει, Για τη μία νομίζουμε έχει ήδη απόφαση κατά της Boeing και αυτό θέτει ένα πολύ σημαντικό προηγούμενο ε, για την βιομηχανία της αεροπορίας σε ό,τι αφορά τις ενισχύσει, Δηλαδή στις 28 Νοεμβρίου το Συμβούλιο ΒΤΟ θεώρησε πως η μαζική χρηματοδότηση για το Boeing 776 αποτελεί παράβαση των κανόνων σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή η χορήγηση των 5,7 δισεκατομμυρίων αποτελεί όχι μόνο παραβίαση, αλλά ουσιαστικά η ε, η κυβέρνηση του, του, του ομόσπονδου της ε, Ουάσιγκτον ε, ε, προέβη και σε αποκλειστική προτίμηση των χωρίως παραγωγμένων τμήματων για το εν λόγω μοντέλο, πράγμα το οποίο επίσης δεν επιτρέπεται. Άρα λοιπόν, εγώ θα πρέπει να πω ότι δεν επιχαίρω ιδιαίτερα αυτό το γεγονό, αλλά ανέφερε ότι WTO ανέφερε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, αντίστοιχα δηλαδή ε, με Λισμπόν και μου είπε ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ε, αλλαγές. Βέβαια το βασικό εδώ πρόβλημα, αν θέλετε, η βασική περίπτωση ήταν αυτή της Μπόν και όχι της Έρμπας. Τώρα σε ό,τι αφορά την Κίνα, μου θέσατε κάποια ερωτήματα. Πέρυσι το Νοέμβριο υπογράψαμε την πλατφόρμα διασυναισιμότητας, το Connectivity ε, Platform, το οποίο θεωρώ πως αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω σχέση μας με την Κίνα. Σε αυτό το τομέα είναι ε, πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ό,τι κάνουμε σε αυτή την ε, πλατφόρμα βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις μας έτσι ώστε να τι αξιώσουμε με το καλύτερο ε, δυνατό ε, τρόπο. Και εδώ αναφερόμαστε ειδικότερα στην διασύνδεση ε, σιδηροδρόμου μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Μετά όμω την πολύ επιτυχημένη σε πολιτικό επίπεδο συνάντηση που έλαβε η χώρα στο Πεκίνο φέτο, τον Ιούνιο, αποφασίσαμε ότι θα ακολουθήσουμε ε, την λογική των διαδρόμων, των corridors, όπως ισχύουν δηλαδή στα διευρωπαϊκά δίκτυα, ώστε να εφαρμόσουμε αυτή την αρχιτεκτονική, αν θέλετε, στον κοινό σχεδιασμό. Και οι δύο πλευρές, και εμείς και η Κίνα δηλαδή, ε, αναφέραμε μία σειρά από project τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο συγχρηματοδότησης και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τα δικά τους ε, project. Λάβαμε λοιπόν έναν κατάλογο έξι project περιλαμβάνονταν εκεί και την τελευταία εβδομάδα λοιπόν παρουσιάστηκε αυτός ο κατάλογος των project ε, στο Πεκίνο και λάβαμε τα πρώτα σχόλια από την πλευρά τους. Άρα λοιπόν εδώ κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και σας είπα ότι αυτό οι διαπραγματεύσει, αυτέ οι συζητήσει υπάγονται στου κανόνε τη ε, κοινή ε, πλατφόρμα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την αμοιβαιότητα. Αλλά αντιλαμβάνομαι και αυτό που είπατε, ότι δηλαδή τα κράτη-μέλη μα θα πρέπει να σέβονται του κοινού κανόνε όταν προμπαίνουμε στη σύναψη συμφωνιών με ε, κοινέου επενδυτέ. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τι δημόσιε προμήθειε, θα πρέπει πραγματικά να τι δημόσιε συμβάσει να ε, δίνονται ίσε ευκαιρίε σε όλες τις επιχειρήσεις για την ε, εφαρμογή των σχετικών project, την εκτέλεση αυτών των project και θα καλέσουμε, να το πω τους ε, κοινούς συναδέλφους να ανταποκριθούν και αυτοί από την πλευρά τους στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δηλαδή, υπήρξε κάποιο πρόβλημα, για παράδειγμα, εκείνη η περίπτωση ε, απόρριψη χρηματοδότηση από την πλευρά τη πολωνικής κυβέρνηση σε σχέση με ένα κινέζικο project. Και να πω ότι και οι δύο πλευρέ ε, συμμετέχουμε στην συνδρομική ε, γραμμή Βουδαπέζης ε, Βελιγραδίου και έχουμε αναφέρει επανειλημμένα ότι σε περίπτωση που υπάρξει εδώ παραβίαση των κοινών κανόνων θα ξεκινήσουμε διαδικασία κατά παράβαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καλωσορίζουμε τους κοινούς επενδυτές. Τους καλωσορίζουμε μεν, αλλά τηρώντας τους εδρεωμένους κανόνες δε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δύο δε. But Αυτό είπατε. Να είμαι ξεκάθαρη στο θέμα αυτό. Και έγινε και μια συνέντευξη τύπου από, μετά το, την απόφαση του Υπουργού Ντόμπριν για το ποια κατεύθυνση θέλει να ακολουθήσει. Να πω ευθύ εξ αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη στην αρχή των διαπραγματεύσεων με τη Γερμανία για την εισαγωγή τέτοιων ε, μηχανισμών επιβολής διοδίων δήλωσε με σαφήνεια τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαμε ενδεχομένω να συμφωνήσουμε και να εγκρίνουμε τέτοιον ε, νομοσχέδιο. Καταρχάς, αναλογικότητα και κατά δεύτερον, ε, μια λύση η οποία θα σήμαινε την κριτική μεταχείριση του οποιοδήποτε. Και εκ παραλλήλου καλέσαμε και τη Γερμανία αλλά και όλα τα υπόλοιπα κρατημέλη γιατί είμαστε υπέρ της αρχής του ορυπαίνων πληρώνει πρόκειται για μια αρχή την οποία ακολουθούμε γενικότερα. Καλέσαμε λοιπόν τα κρατημέλη να ακολουθήσουν την αρχή αυτή. Καλέσαμε επίση τη Γερμανία να λάβει υπόψη ναι, και τη ε, ε, επιβολή διοδίων ανά απόσταση. Αυτό όμω δεν είναι νόμος, αυτό ήταν απλά μια σύσταση. Αναζητούμε μια πανευρωπαϊκή λύση και αυτό ασφαλώς αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων και στο Συμβούλιο. Αυτό θα περιλάμβει και η πρότασή μας του χρόνου. Εκεί λοιπόν εστιαστήκαμε με συνέπεια. Και όντως ο πρόεδρος Γιούγκερ μίλησε με Γερμανούς αντιπροσώπους, ε, αλλά υποστήριξε ακριβώς τα σχέδια αυτά. Ποτέ δεν ε, έπεσε επιτάπητος οποιαδήποτε άλλη λύση. Πάντα λοιπόν με αναλογικότητα και με διακριτική μεταχείριση. Τι πετύχαμε τώρα. Τι πετύχαμε και γιατί υποστηρίζουμε την πρόταση. Καταρχάς, η Γερμανία πληρεί τον όρο της αναλογικότητας σε ό,τι αφορά την επιβολή ιδιωδίων. Είμαστε τώρα στο 2,5 ευρώ ανά, ανά 10 ημέρες, το οποίο είναι αναλογικό με το ετήσιο σήμα το μπινιέτ. Κατά δεύτερον, η Γερμανία έχει γενικώ δικαίωμα να επιβάλλει τέλη, όπως επιβάλλουν τέλη και πολλά άλλα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο που πετύχαμε και αυτό ήταν σημαντικό. Να κατανοήσετε ότι δεν μπορούμε να αναμειχθούμε παντού, αλλά μπορούμε να αναμειχθούμε στο πώς υπολογίζεται το ποσό που επιβάλλεται αποσυνδέθηκε το ποσό αυτό από τα τέλη τα οδικά. Αυτά είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Δεν μπορώ να αποφασίσω όμως και να παρέμβω στο πώς επιβάλλει φόρους η Γερμανία. Αυτό είναι αντικείμενο άλλες συζήτηση. Στην παρούσα φάση οι οδικές, τα τέλη, τα οποία αποτελούν αντικείμενο των νόμων για τις μεταφορές έχουν αποσυνδεθεί και από την πρώτη ημέρα το ζητούσε αυτό και πολεμούσε γι' αυτό. Άρα, ό,τι και να γίνει στο μέλλον για τις οδικές μεταφορές, αυτό θα είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες, δύο διαφορετικοί φόροι και γι' αυτό εγώ είμαι ικανοποιημένη. Αλλά στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ακόμα το αναθεωρημένο μοντέλο για την Ευρώπη. Και τα λάβατε και την πρότασή μας τον Απρίλιο του χρόνου, ελπίζουμε. Αυτό είναι ο στόχος μου. Θα υπάρχει ηλεκτρονική επιβολή λοιπόν τελών, οδικών τελών, ε, διοδίων και το θέμα του σήματος οδήγησης. Αλλά να πω επίσης ότι δεν έχουμε ακόμα εγκρίνει το οτιδήποτε, γιατί φυσικά πρώτα θα πρέπει να δούμε το νομοσχέδιο το οποίο θα δημοσιευθεί στην επίσημη γερμανική εφημερίδα και μόνο τότε θα μπορούμε πραγματικά να αποφασίσουμε στην παρούσα φάση το μόνο που κάναμε είναι να βάλουμε σε πάυση όλη τη διαδικασία μέχρι ότου δούμε την επίσημη πρόταση νομοσχεδίου της Γερμανίας για τον 868. Ε, Ένα μισή χρόνο μόνο το δουλεύουμε. Και συμφωνώ ότι δεν είμαστε και ταχύτατοι. Όλοι θα το θέλαμε πιο γρήγορα, αλλά 868 είναι ένα από τα εργαλεία στο πακέτο των διαπραγματεύσεων για την αεροπλοεία. Είναι ένα εργαλείο του πακέτου. Δεν είναι τμήμα τη συνοπτική ε, συμφωνία. Είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσει η συνοπτική συμφωνία. Άρα, μετά το νέο έτος με το καλό, ελπίζω να είναι έτοιμη η πρόταση αυτή για να την ε, λάβατε κι εσείς. Εγώ το προωθώ ιδιαίτερως αυτό. Πρώτα και καλύτερα, γιατί το χρειάζομαι το εργαλείο αυτό. Ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσει. δεν ήταν απαραίτητο κατεπήγον να το έχουμε στην πρώτη φάση, γιατί είναι ένα από τα θέματα που θα κοιτάξουμε τελευταία, αλλά το θέλω, οπωσδήποτε στην εργαλειοθήκη μου. Και τώρα να περάσω. Μήπως δεν έχω και χρόνο, δεν ξέρω. Ένα πράγμα μου θέλω να πω, ένα πράγμα το οποίο όλοι σας, ή τουλάχιστον πιο πολύ το δείξατε, το πακέτο για τις οδικές μεταφορές. Λίγο συνεπτικές πληροφορίες επιτρέψτε μου να σας δώσω, κυρίως για κοινωνικά ζητήματα. Καταρχάς, εγώ θέλω για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα, forum shipping, καμπότας, ελάχιστη μισθή, όλα αυτά τα θέματα θέλω να υπάρχουν πανευρωπαϊκές λύσεις, πανευρωπαϊκές λύσεις αναλογικές που να συνάπτουν με την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, όπως σας είπα. Για να δούμε λοιπόν τα θέματα αυτά. Το Forum Shipping, Letterbox Companies, ε, ε, δηλαδή εταιρείε γραμματοθρίδας. Εδώ θα πρέπει οι εταιρείες να καταχωρίζονται εκεί όπου διεξαγάγεται η πλειονότητα των επιχειρήσεων και των συναλλαγών τη επιχειρήση. Ελπίζω να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Ένα άλλο θέμα. Η καλή φήμη. Θέλουμε να προωθήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών. Για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα καλύπτεται μόνο η ασφάλεια στους δρόμους στην ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και όλη η κοινωνική κανόνες και αυτοί θα αποτελούν τμήμα της ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό προτείνουμε. προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους ε, παράγοντες που παρουσιάζουν προβλήματα και να τους αντιμετωπίσουμε για να δημιουργήσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για το καμποτάζ. Δεν προγραμματίζουμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά εκ βάθρων. Θέλουμε απλά να εξασφαλίσουμε να υπάρχουν ε, κοινέ εξηγήσει των υφιστάμενων νόμων και να είναι εφαρμόσιμε. Προ αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα κινηθούμε. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπήρξε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Αντί να μετρήσουμε τον αριθμό των pickups στην επιστροφή, να συζητάμε την απόσταση και το χρονικό περιθώριο το οποίο έχει το φορτηγό για να βγει από τη χώρα. Και φυσικά συναντιέμαι, ε, θα συναντηθώ μάλλον με εκπροσώπους των ενώσεων ε, των ε, οδηγών φορτηγών των Ιανουάριο στις Βρυξέλλες για να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος για τον ελάχιστο μισθό τώρα, τον κατώτατο. Εδώ έχουμε σοβαρές προκλήσεις γιατί οι κατώτατοι μισθοί ε, διαιρούν φυσικά και τεχάζουν τον την Ευρώπη και υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα και από τους μεν και από τους δε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό συμφέρον το να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση. και μετά την οδηγία για του single workers θα πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση για τι μεταφορέ. Δεν μπορεί να ισχύουν οι ίδιε οι κανόνε. Και χαίρομαι που είναι συμφωνεί ο συνάδελφο Τέισεν. Η συνάδελφο Τέισεν. Θα υπάρχει ιδιαίτερη μνήμα σε ό,τι αφορά τους ε, εργαζόμενου που χρησιμοποιούν τι μεταφορέ αυτέ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ειδική πρόταση. Δεν νομίζω ότι αρκούν αυτά που έχουμε επιτάπητο στην παρούσα φάση. Θα πρέπει να πάμε και λίγο παραπέρα, να βρούμε κάτι το οποίο θα απαντήσει στι ανησυχίε και των δύο πλευρών. Και αυτό που θα ήθελα εδώ να επισημάνω για το θέμα αυτό, σας παρακαλώ να αποφύγουμε τον καταγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Γιατί αν επιτρέψουμε τον καταγραμματισμό, θα το τέλος της Ενιαίας Αγοράς. Και αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτός είναι ο απότερος στόχος μου και θα συνεχίσω ανελειπώς να καλώ όλους τους φορείς να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις απάτες και τις, ε, το πείραγμα των ταχογράφων. Έγινε διάφορα τα σχόλια και θα προβούμε και σε νέες τεχνικές προδιαγραφέ σε ό,τι αφορά τους ταχογράφους. Αν τα κρατημέλη και το Συμβούλιο είναι βιτεθειμένα να κινηθούν πιο γρήγορα, ευχαρίστω. Εγώ πρώτα και καλύτερη. Αλήθεια, σας το λέω. Έχουμε καινούργια τεχνολογία. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αν θέλουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά πιο γρήγορα, πολύ ευχαριστώ. Άλλο θέμα το οποίο και αυτό θα μπει μάλλον στο πακέτο. Το ακούμε όλο και πιο συχνά στα σχόλια των κρατών μελών. σε ό,τι φέρνει τα φορτηγά κάτω από 3,5 τόνου. Γιατί από ό,τι φαίνεται και εκεί είναι μεγάλε οι απάτε και ζήτησα από τα κράτη-μέλη να μου δώσουν ε, αποδεκτικά στοιχεία, τεκμήρια, για να τι εξετάσουμε από πλευρά τη υπηρεσία. Στην παρούσα φάση όμω δεν έχω κάτι σίγουρο, μόνο φήμε. says to plus. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αλλά είναι γεγονός, όπως ξέρετε και εσείς όλοι σας, ότι είναι θέμα επικουρικότητας. Είναι θέμα επικυριαρχίας δύο κρατών μελών. Εμείς χρησιμοποιήσαμε και εξαντλήσαμε όλα τα διπλωματικά μέσα. Είμαι απογοητευμένη δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοια τοποθέτηση στην ευρωπαϊκή πολιτική. Καλό. Την Ισπανία και την ε, Αγγλία. Να μετακινηθούν για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Δεν έχει νομικά μέσα στα χέρια της Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δεμένα τα χέρια μας. Είναι μεταξύ Ισπανίας και Μεγάλης Βρετανίας. Σας καλώ όλους σας. Κάντε ό,τι μπορείτε. για να υποστηριχθεί με κάποιο επικοδομητικό τρόπο αυτό ο διάλογο και να βρεθεί μια λύση. Γιατί όλη η αεροπλοεία διακυβεύεται. χάζουμε και δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια σα λέω. Επειδή δεν υπάρχει ε, αποτελεσματικότητα στο Single European Skies. Ενώ υπάρχουν λύσει. Υπάρχουν λύσει. Δεν ξέρω. Ίσως ε, μια επόμενη γενιά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ απογοητευτικό πάντω και χρειάζονται νέε λύσει. Δεν ξέρω. Ήλπιζα για ένα θετικό αποτέλεσμα, μια θετική εκβάση. Δεν έχω χάσει την τελευταία μου ελπίδα. Uber. Όπως είπατε, στην περίπτωση της Uber. Πιστεύω ότι τελικά το ψήφισμα κινείται προ την κατεύθυνση ότι να ορίζει η εθνική νομοθεσία, ε, αν πρόκειται για δημόσια συγκοινωνία ή όχι. Κατά πάσα πιθανότητα χρειάζεται πανευρωπαϊκή υπηρεσία, αλλά κοιτάξτε, οι υπηρεσίε ταξί είναι αστικέ ε, ε, υπηρεσίες. Εμάς μας απασχολούν πιο πολύ τα διασυνοριακά στοιχεία τη των μεταφορών. Προ την κατεύθυνση λοιπόν αυτή θα συνεχίσουμε να, βρίσουμε, να κάνουμε διάλογο για να βρούμε μια λύση. Έχω δύο ανησυχίες, ανησυχίες σε ό,τι αφορά τη συνεργατική οικονομία, όχι τόσο την Uber. Ανησυχώ λοιπόν, γιατί πιστεύω ότι προωθούμε την κατάργηση των ε, τοπικών μονοπωλίων, αλλά δημιουργούμε παγκόσμια μονοπόλια από δίπλα ακριβώ παράλληλα. Και δύο στοιχεία. Ο συνάδελφος Μοσκοβισή προσπαθεί να επιβάλλει την αρχή επιβολή των φόρων εκεί που ε, γίνεται και προκύπτει το κέρδο. Αυτό είναι βασικό και θα μας βοηθούσε πολύ. Η δεύτερη ανησυχία μου είναι τι θα συμβεί στο εργατικό δυναμικό, γιατί είναι τεράστια τα αριθμητικά στοιχεία στην συνεργατική αυτή οικονομία. Άμα ξαναλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο και αυτός ο κόσμος μείνει τελικά στον αέρα, χωρίς κάποια συγκεκριμένη κατάρτιση, εκπαίδευση, διαβίου τα κτλ. Αυτέ είναι οι ανησυχίε μου, δύο από τι ανησυχίε μου. Θα συνεχίσουμε να τα εξετάζουμε τα θέματα αυτά, θα πρέπει να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις και πάλι. Όχι τόσο για την Uber, αλλά για τη συνεργατική οικονομία εν γέννη. Για τους ε, στόχους. Να σας δώσω σύντομα κάποια στοιχεία για την οδική ασφάλεια. Άλλος ένας τομέας απογοήτευσης. Αλλά όλοι οι φορείς, οι υπηρεσίες μου, όλοι συνεργαζόμαστε και θα βρούμε μια λύση, είμαι σίγουρη. Είχαμε 135.000 σοβαρούς τραυματισμούς ετησίως στην Ευρώπη. Φανταστείτε έτσι, 135.000 σοβαρούς τραυματισμούς ετησίω στην Ευρώπη. Φανταστείτε πόσες οικογένειες εμπλέκονται εδώ, σοβαρά. 26.000 θύματα επίσης ετησίω. ετησίως. 26.000 θύματα ετησίως. Σοβαρά στοιχεία αυτά. Και ναι, αγαπητέ Βαντερκάπ, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πετύχαμε τίποτα. Ναι, έχουμε τα στοιχεία, αλλά δεν προχωράμε. Για να φτάσουμε στους στόχους του 2020, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί το πρόβλημα είναι τώρα ότι ακόμα και οι πιο επιτυχείς χώρες έχουν αδρανίσει. Και με το CITS είχα ελπίδες ότι θα έχουμε νέες λειτουργίες με τα αυτοκίνητα που θα αυξήσουν τις δυνατότητες δημοσίων ή πολυτροπικών μεταφορών. Έχουμε ψηφιοποίηση η χώρα παντού, σε όλο το τομέα των μεταφορών. Και βέβαια, του χρόνου θα τα ανακοινώσουμε όλα αυτά βάσει της επερχόμενης έκθεσης για τους σοβαρούς τραυματισμούς. Θα ανακοινώσουμε και τους στόχους Νομίζω 16 χώρες μέλη μας δίνουν στοιχεία για σοβαρούς τραυματισμούς. Καλό όλους λοιπόν τους υπουργού, όλα τα υπουργεία να, να μας στείλουν στοιχεία μέχρι το Μάρτιο του χρόνου, ώστε τουλάχιστον να έχουμε ένα μοντέλο κατά προσέγγιση μέσα στα πλαίσια του οποίου μετά να θέσουμε σοβαρούς ε, στόχους για τους τραυματισμούς σοβαρούς. Επίσης, υπό Μαλτίζικη Προεδρία και υπό την αιγίδα του Άτυπου Συμβουλίου θα κάνουμε μια παγκόσμια διάσκεψη για την οδική ασφάλεια σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και τους πρεσβιστού και θα χαρώ πολύ για την πιθανή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Είχαμε θετικά αποτελεσμάτα πάντως. Η Πολωνία, α πούμε, βελτίωσε τι στατιστικές τη μαζί με 23 φορεί προσπάθησαν να κάνουν ολιστικό μοντέλο και ξέρω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά μετά από πολλή προσπάθεια βέβαια και συντονισμό τα οποία είναι απαραίτητα για να προχωρήσει κανείς το Edward είναι επίσης πολύ ενθαρρυντικό γιατί θέλουμε να φτάσουμε μια μέρα χωρίς θύματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους και είχαμε πετύχει μια συγκεκριμένη μέρα πραγματικά στο σχεδόν εκμεδενισμό των σοβαρών ατυχημάτων και των θανάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Θα σταματήσω εδώ, ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά πολύ ευχαριστώ να απαντήσω σε όποιους επέβαλαν ερωτήματα άμεσα και δημερώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και Πρόεδρος. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε ταχύτατα τα κλεισμένο των θυρών. Επόμενη συνεδρίαση 25 Ιανουαρίου του 2017 στις 9 το πρωί. Συνεχίζουμε λοιπόν και κλεισμένων των θερών. Είναι ουσιαστικά για τους συντονιστές αυτή τη συνεδρία, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν και μέλη της Επιτροπής. Ωστόσο, όχι το κοινό. Οπότε, αποχωρήσει το κοινό τώρα από την αίθουσα και θα συνεχίσουμε μετά με την έκθεση από το της Επιτρόπου σε ό,τι